Κοινοβούλιο μετά τις πρώτες εκλο... άμεσες εκλογές. Ε, αυτό είναι αλήθεια και καλό είναι να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, θα ευχαριστώ πολύ που μου ανατέθηκε η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κλείνει εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30. Τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε τη δήλωση της ύπαρξης εκπροσώπου ε, σχετικά με την κατάσταση στο Μαλί. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Στις 21 Μαρτίου έγινε πραξικόπημα στο Μαλί που ξεκίνησε από μια εξέγερση του στρατού που ζητούσε καλύτερα όπλα και καλύτερη ε, ε, ηγεσία ε, από την εξέγερση που κινήθηκε προς τα βόρεια. Η Έκουβα, η οικονομική κοινότητα των χωρών τη Δυτική Αφρική συνεχίζει να ασκεί πίεση μαζί με τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, πιέζοντα προ μια ε, συμφωνία που ε, στις στι 6 Απριλίου για επιστροφή σε μια μη στρατιωτική κυβέρνηση. Ε, εν τω μεταξύ, ορίστηκε ένα ε, ε προσωρινό πρόεδρο, ο Διοκούντα Τραωρέ, και οι εκλογέ ε, θα πρέπει να διεξαχθούν αμέσω μόλι ολοκληρωθεί η ολοκληρωθούν ε, οι εκλογικοί κατάλογοι. Η κατάσταση αυτή επιδίνωσε πάρα πολύ ε, την ε, κατάσταση στο βόρειο Μαλή όπου οι αντάρτες κατάλαβαν τρεις πόλεις μεταξύ των οποίων και το Τιμπουκτού οι Τουαρέγ ανακήρυξαν την ανεξαρτησία σε μια περιοχή εκεί που εμέσως απορρίφθηκε από την Ένωση, την Βόρειο Αφρικανική Ένωση ε, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για την ευαλωτότητα του Σαχέλ εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Γίνεται όλο και πιο σαφέ ότι η ανάπτυξη και η ασφάλεια πρέπει να προχωρήσουν ε, παράλληλα. Ε, έτσι προτείνουμε μια συνολική προσέγγιση ε, μέσω μια στρατηγικής για το Σαχέλ που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο πριν από ένα χρόνο και διορίστηκε έτσι ένα ανώτατος συντονιστή για το Σαχέλ. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μια πρόσθετη χρηματοδότηση 50 εκατομμυρίων έδωσαν συμβολή στην υποστήριξη τη πολιτική ασφάλεια του Μαλή. Η κρίση στη Λιβύη και οι επιπτώσει τη επιδίνωσαν ένα ήδη υπάρχουν πρόβλημα ε, ε, καθώς ε, οπλισμένοι μαχητές πέρασαν στην περιοχή αυτή όπου η τρομοκρατία, οι ομοιρίες, η λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η εγκληματικότητα ήταν ήδη σοβαρά προβλήματα. Ε, μαζί με την συνεχή ανασφάλεια όσον αφορά τα τρόφιμα, μια μείζων διατροφική κρίση επιδίνωσε σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Ε, έχω ε, έρθει σε επαφή ε, και μάλλον γενικά όταν οι κυβερνήσει στην περιοχή αυτή είναι ισχυρέ, η κατάσταση είναι καλή. Αλλά το ε, στρατιωτικό πραξικόπημα στο Μαλί ε, τέλειω υπονόμευσε και την νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα τη κυβέρνηση. Ε, καταδικάστηκε ε, το πραξικόπημα στις 22 Μαρτίου και ζητήσαμε ε, την αποκατάσταση μιας νόμιμης δημοκρατικής κυβέρνησης και διεξογείου εκλογών. Στις 23 Μαρτίου το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υποστήριξε τις προσπάθειες της οικονομικής κοινότητας των χωρών της Δυτικής Αφρικής, ΕΚΟΒΟΑΣ, για την αποκατάσταση συνταγματικής και δημοκρατικής κυβέρνησης στη Μαλή. Ε, κάθε αναπτυξιακή συμφωνία που είχαμε και συνεργασία με την κυβέρνηση του Μαλή αμέσως αναστάλθηκε με το πραξικόπημα, αλλά αυτό δεν επηρέασε οποιαδήποτε άμεση βοήθεια προς τον λαό. Χάρη στην διαμεσολάβηση της ε, Πουρκίνα Φάσο, στις 6 Απριλίου επετέχθη συμφωνία με τους στρατιωτικούς που δεσμεύει όλα τα μέρη και τους ε, στρατιωτικούς να ε, υπάρξει πλήρη σεβασμός ε, και αποκατάσταση της δημοκρατικής ε, διακυβέρνησης. Ε, μίλησε στις 7 Απριλίου στον πρόεδρο Οατάρα, πρόεδρο του, της με σκοπό να ενισχύσω αυτό το μήνυμα. Ε, και με τον Μπάκι Μουν μίλησα χθε για το θέμα αυτό στις Βρυξέλλε. Η ανάλυση καθηκόντων από τον Διορκούντα Τραωρέ ως ε, προσωρινού Προέδρου και η απελευθέρωση των κρατούμενων υπουργών ήταν ε, καλά νέα. παρόλο που οι συλλήψει άλλων πολιτικών και στρατιωτικών προκαλεί μεγάλε ανησυχίε και θα είναι στην ημέρια διάταξη την επόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο Εξωτερικών. Ε, μόλις ε, ε, λειτουργήσει η προσωρινή κυβέρνηση θα αρχίσουμε να συζητάμε μαζί τους σχετικά με την ε, μεταβατική περίοδο και την ε, διεξαγωγή εκλογών μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ελπίζουμε ότι η πλήρη τήρηση τη συμφωνία με την ΕΚΟΒΟΑΣ θα οδηγήσει στην υποκατάσταση μια δημοκρατική και νόμιμη κυβέρνηση. Ε, θα δώσουμε όποια υποστήριξη ε, χρειάζεται η κυβέρνηση από του εξωτερικού εταίρου και αυτοί θα αποφασίσουν τι και από ποιον. Ε, θα φροντίσουμε για τον τομέα τη ασφάλεια, ιδίω στα βόρεια τη χώρα, σε στενή συνεργασία με τι τι χώρε, χώρε, Μαυριτανία, Νίγηρα, Αλγερία, Μπουργίνα Φάσο και Ακτή Ελεφαντοστού. Όλε οι χώρε αυτέ έχουν ε, σαφώ ε, μεγάλο ενδιαφέρον για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο Μαλί. Ε, κάτι τέτοιο δείχνει ε, ποια θα μπορούσε να είναι η φύση μια τέτοια αποστολή και πώ ε, θα πρέπει, πόσο απαραίτητο θα είναι ο συντονισμό και η ενίσχυση και του Εθνικού Στρατού και τη χωροφυλακή του Μαλί. Ήδη στι 21 Μαρτίου, την, την ημέρα δηλαδή του πραξικοπήματο, οι συμπρόεδροι τη Κοινοβουλευτική Επι... Ε, Συνέλευση ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν την ε, βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση στην κατάσταση ε, στο Βορρά. Το Συμβούλιο ξεκαθάρισε την προσήλωσή του στην εδαφική ακαιρεότητα του Μαλή και την ανάγκη να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η δημοκρατία στον Βορρά. Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επίγουσα λόγω τη της ε, μεγάλης ανθρωπιστικής ε, κρίσης. Ε, συνολικά πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά στο Μαλί, ενώ πάνω από 140.000 εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει σε γειτονικέ χώρες. Για το 2012 αυξήσαμε τον προϋπολογισμό μας για την ανθρωπιστική βοήθεια προς το Σαχέλ από 45 εκατομμύρια σε 105 εκατομμύρια ευρώ. για την Μαυριτανία, Νίγηρα, Τσάντ, Μαλί και Μπουρκίνα Βάσο, η Κομισιόν χρησιμοποιεί πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια και δράσει για την διατροφική ασφάλεια για έναν εκτιμόμενο πληθυσμό 50 εκατομμυρίων ανθρώπων. Επιπλέον 9 εκατομμύρια προστέθηκαν νωρίτερα το μήνα αυτό για τρόφιμα, καταφύγια και ε, νερό για τους πρόσφυγες από το Μαλί και τους εσωτερικά εκτοπισμένους. Ε, αυτή τη στιγμή ο πρωτοαρχικός μας στόχος είναι ε, να προσφέρουμε μέσα άμεσης ανακούφισης για, τους πιο, ε, για τα πιο ευάλωτα μέρη του πληθυσμού. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με τις νέες προσωρινές αρχές στο Μπαμάκο με σκοπό να προσδιοριστεί τι συγκεκριμένη βοήθεια θα μπορέσουμε να δώσουμε σε επίπεδο τροφίμων, ε, εκλογικής διαδικασίας, ε, ασφάλεια κλπ. Η σταθερότητα στην περιοχή αυτή είναι θεμελιώδη σημασία για όλη αυτή την περιοχή της Αφρικής και γι' αυτό έχουμε σε σκοπό να κινητοποιήσουμε όλες μας τις προσπάθειες προσπάθειες για να βρεθούν λύσεις όχι μόνο για τα επίγοντα προβλήματα των επόμενων εβδομάδων αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Με τη σαφή μας πρόθεση να βοηθήσουμε το Μαλί να ανακτήσει την ε, κυριαρχία του στο βόρειο μέρος της χώρας και να γίνει πραγματικά ένα ενωμένο έθνος. Σα ευχαριστούμε, κυρία είπατε την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα εισαγωγικά σα σχόλια. Τώρα θα περάσουμε στους ομιλητές. Ο κύριος Κασουλίδης πρώτα για δύο λεπτά από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόσφατο πραξικόπημα στο Μαλί επισημαίνει το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν αυτόν τον καιρό περιφερειακές αφρικανικές οργανώσεις, εν προκειμένου η ΕΚΟΒΑΣ, η Οικονομική Κοινότητα δικοαφρικανικών Χωρών, σε ό,τι αφορά την άσκηση πίεσης για αποκατάσταση της συνταγματική τάξης και της κοινοβουλευτική πλουραλιστική δημοκρατία. Τα πραξικοπήματα δεν γίνουν πλέον αποδεκτά από τις ίδιε τι αφρικανικές χώρες. Παρόμοιο ρόλο ε, διαδραμάτισε η ΕΚΟΒΑΣ και για την ακτή του ελεφαντοστού. Βέβαια, ιδιαίτερα ε, προβληματική όχι μόνο για την Αφρική αλλά και για την ε, ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη είναι η εξελίξη στο Βόρειο Μαλί, γιατί έχουμε ε, ένοπλους μαχητές που ε, ήταν μισθοφόροι του Καντάφη και ισλαμιστικά ακρεφνή ε, εξεμιστικά κινήματα που υποστηρίζονται από την Αλκάιντα και το Μαγκρέμπ εκμεταλλεύονται την κατάσταση και εξασφάλισαν την επικράτησή τους σε χώρες όπως το Κιντάολ του Μποκτού και μάλιστα μονομερώς εν, ανακήρυξαν την ανεξαρτησία του κρατού Σαββάμπ. Τέτοιες αναγνωρίσεις τέτοιες ανακηρύξεις μετατρέπουν ορισμένες περιοχές σε καταφύγια για τρομοκράτες και θα δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη την περιοχή του Σαχέλ, όχι μόνο στη, στο Μαλία, στη Μαυριτανία, στον Ήγυρα, στον Μπουρκίνα Φάσο. Είναι γνωστή άλλωστε αυτή η περιοχή για απαγωγές και ανομία και από το παρελθόν. Θα πρέπει να διατρανώσουμε την υποστήριξή μας για την εδαφική ακαιρεότητα και την ενότητα του Μαλή. Οποιαδήποτε απόσχεση, απόσχεση ε, ε, τμήματος της επικράτειας είναι απαράδεκτη. Θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε τον συνταγματικό πρόεδρο, τον Ντίον Κούντα Τραωρέ και χαίρομαι ιδιαίτερος κυρία είπατε εκπρόσωπε που το διευκρινίσατε αυτό γιατί είναι σημαντικό για την ε, επαναφορά και αποκατάσταση της εδαφικής ε, ενότητας και καιρότητας του Μαλή. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη μεγάλη καθυστέρηση, γι' αυτό θα πρέπει να τηρούμε πολύ πιστά το χρόνο μας. Για ένα λεπτό, κυρία Γκόμες, είναι η επόμενη η Δεν είχαμε δεν είχε σταματήσει ο απόϊχος του πραξικοπήματος στο Μαλί και ξεκίνησε, ακούσαμε τα νέα για το πραξικόπημα στη Γουινέα Μπισάου. Δύο πραξικοπήματα μέσα σε δύο εβδομάδες. Θα πρέπει να δούμε τη σχέση μας με την ΕΚΟΒΑΣ, με την ε, Οικονομική Κοινότητα Δυτικοευρωπαϊκών Χωρών, με την ΑΚΕ και κυρίως να σταθεροποιήσουμε πληθυσμούς που χρειάζονται δημοκρατία, κράτος δικαίου και σταθερότητα για να αναπτυχθούν. Ε, αυτό ενδιαφέρει και την Ευρώπη και τη σταθερότητά τους γιατί ε, από τις χώρες αυτές παίρνουν ναρκωτικά, όπλα που κατευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε μηχανισμούς για να αντιδράσουμε στην κατάσταση αυτή. Δεν αρκούν ε, κάποιες διακηρύξεις ε, και καταδίκες. Θα πρέπει να τις συνδυάσουμε με διπλωματική προσπάθεια και με την χρήση της ΕΠΑ και τη χρήση της επισητιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει μπροστά στις απειλές αυτές να υψώσουμε τη φωνή μας και να αντιδράσουμε. Ήταν απαράδεκτο το κλείσιμο της αποστολής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη, διακόπτεται το μικρόφωνο της uh, κυρίας Γκόμες. Λυπούμε, λέει ο πρόεδρος, εγώ σας διακόψα κυρία Γκόμες, γιατί όπως είπα και προηγουμένως έχουμε σημαντική καθυστέρηση και επίσης θα ήθελα να ζητήσω από τους να μιλούν πιο αργά για να μπορούν να του παρακολουθούν και οι διερμηνείς. Ήταν ε, πραγματικά μεγάλη ταχύτητα με την οποία μιλούσε η κυρία Γκόμες. Ο κύριο Γκέρνη, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το τι κρίμα. Έχουμε μία κρίση, ε, έχουμε κρίση μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια ήταν πρότυπο δημοκρατίας ε, και σταθερότητας. Το Μαλί θα πρέπει να αντιμετωπίσει ε, πολλέ προκλήσεις. Καταρχήν, ε, παραφορά του κρατού δικαίου, της εδαφική ε, ακαιρεότητα και εξασφάλιση της ευημερία των πολιτών που αυτή τη στιγμή εξαρτούνται από την εξωτερική ενίσχυση. Πώς αντιμετωπίσει αυτές τις τρεις προκλήσεις το Μαλί. Βέβαια, τι ίδιε απειλέ αντιμετωπίζουν και γειτονικέ χώρε. Οπότε η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί, η αντίδραση θα πρέπει να είναι περιφερειακή. Γι' αυτό και είναι θεμελιώδη ο ρόλο ε, τη ΕΚΟΒΑΣ που έχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω Ευρωπαίοι έχουμε ένα προφανέ ε, συμφέρον και ενδιαφέρον να βοηθήσουμε την ΕΚΟΒΑΣ και να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική που θα εφαρμόσουμε στη μετά τον κατάφη εποχή γιατί εν μέρη τα γεγονότα στη Λιβύη ξεκίνησαν από τις γενικότερες εξελίξεις στη ζώνη του Σαχέλ. Έχουμε πολύ πλούσια πείρα αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες αυτές. Θα πρέπει να τρίσουμε διδάγματα από την βοήθεια αυτή. Πριν από ένα χρόνο είπαμε ότι η στρατηγική μας στη ζώνη Σαχέλ θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Θα πρέπει η κατάσταση φυσικά να επανέλθει σε ένα ψυχολογικό δρόμο το συντομότερο δυνατό για να συνεχιστεί η αναπτυξιακή βοήθεια που ανεστάλλει μετά το πραξικόπημα στο Μαλί. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που τηρήσατε και το χρόνο σας. Η επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Σαρτζεντίνη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από δύο εβδομάδες πήγα στο Ισενεγάλη, στο Ντακάρ και είδα του Αρέγκ που είχαν διαφύγει από το Ομαλή ήταν ένας του Αρέκ πολύ καλός και μορφωμένος άνθρωπος ε, με ανοιχτό πνεύμα τα παιδιά του, αγόρια και κορίτσια, είχαν πάει στο σχολείο, είχαν σπουδάσει, αλλά δεν ζούσαν στο Μαλί επειδή ήταν επικίνδυνο και ο του Αρέγ φοβόταν τις διακρίσεις. Ε, τους ε, ε, αντιμετωπίζουν ε, προσχηματικά μιλούν για το Ισλάμ και πολλοί όμως δεν έχουν μπει ποτέ σε ένα τζαμί το, τα μηνύματα αυτά λοιπόν είναι επικίνδυνα. Όταν έφυγα από τον Τουαρέγ δεν είχα καταλάβει ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημα. Κατάλαβα όμως ότι στο Μαλί δεν πρόκειται για μια σύγκρουση καινούρια που τώρα μόλις άρχισε. Υπήρχε έλλειψη συνεργασίας, έλλειψη αμοιβαίου σεβασμού εδώ και γενναίες πίσω. Και τώρα ε, για άλλη μια φορά βλέπουμε την άνηση κατανομή του πλούτου. Υπάρχει ε, πλούτο στο Μαλί, ε, πλούσιο υπέδαφος, αλλά δεν χρησιμοποιείται σωστά και δεν κατανέμονται τα κέρδη δίκαια. Ευχαριστώ. Ο ευχαριστώ. Βεβαίως ε, καταδικάζομαι την ε, ε, δήλωση ανεξαρτησίας του Αζαβουάντ το οποίο ανέφερε και ο πρόεδρος τώρα. Τώρα θα πρέπει οι βόρειες περιοχές να δεθούν υπό έλεγχο από τις κεντρικές πολιτικές αρχές. Οτιδήποτε άλλο θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή Σαχέλ που είναι πολύ σημαντική. Ε, το MNLA, ε, το Εθνικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Ασαβάντα, θα πρέπει να συμβιβαστεί είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι εξτρεμιστές, ε, οι μέλη της Ακάιντα ε, χρησιμοποιούν πολύ βίαιες ε, μεθόδους, απαγωγές μεταξύ άλλων. Είπα ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ενωσιακά κονδύλια ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα του Μαλή ε, ούτως ώστε να μπορέσει ε, και μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών με τον καινούριο πρόεδρο να οδηγηθούν σε σταθεροποίηση και δίκαιες εκλογέ. Για 1,5 λεπτό τώρα, κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το Μαλί και για τους καημένους τους Μαλίαν, για τους κατοίκους του Μαλή, για όσους ζουν σε μια περιοχή του κόσμου που αντιμετωπίζει μια υγειονομική και ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου, που όπως είπατε και εσείς κύριε Άστον, δεν ξεκίνησε με τη νέα εξέγερση το προηγούμενο Ιανουάριο, ούτε με την ανταρσία της 21ης Μαρτίου. Ε, το Μαλί αγνοήθηκε στην προσπάθεια αποικιοποίησης και η Γαλλία φέρει βαρύτατες ευθύνες για την κατάσταση αυτή. Σπάνια τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που δόθηκαν στους Τουαρέγκ. Στην ε, περιοχή αυτή είναι πολύ σημαντικές οι βλέψεις εξαιτία του σημαντικού ορυκτού πλούτου και των φυσικών πόρων και μάλιστα όχι από τις γειτονικέ μόνο χώρες αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες. Πάνω από 10 χρόνια η ζώνη Σαχέλ είναι μια ζώνη στην οποία ανθεί το χειρότερο λαθρεμπόριο χωρίς κανένα έλεγχο και με πλήρη ανομία. Μετά το τέλος του πολέμου της Λιβύης ε, είχαμε εισαγωγή λαθρεμπόριο όπλων στο Μαλή και μετά τον αφοπλισμό των αντάρτων της Λιβύης οπλίστηκαν οι αντάρτες του Μαλή και έχουμε κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδιαίτερα των γυναικών. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήψει το ε, Μαλή, αλλά να κάνει ένα απολογισμό των κονδυλίων που έχει ήδη αφιερώσει τη χώρα αυτή και που δυστυχώς δεν φτάνει στους ε, άμεσους δικαιούχους που είναι οι πολίτες. Θα πρέπει να διαλευκανθούν όλες οι καταχρήσεις και όλες οι παρανομίες ε, που έγιναν θα πρέπει να ε, στηριχθεί μια πολιτική λύση με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, ακόμη και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Γκάλερ. Κυρίες και, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι στην πολιτική αξιολόγηση της κατάστασης στο Μαλί συμφωνούμε όλοι. Και Χαιρόμαστε διότι οι εξελίξεις πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την πρωτεύουσα τουλάχιστον την ε, πρωτεύουσα και το περίγυρό της το πρόβλημα της κατοχής ε, ε, βέβαια και της μονοπλευρής δήλωσης ανεξαρτησίας δεν έχουν λυθεί. Εμείς μπορούμε να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει λοιπόν να αποσταλεί και πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρονικό αυτό διάστημα για να φροντίσουμε ώστε η ECOWAS, το Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Χωρών, να αναλάβει δράση. Ήδη υπάρχει ε, προηγούμενη ε, ε, εμπειρία ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι ότι αρχίζοντας από τη Δυτική Σαχάρα, Μαυρετανία, Νίγερα, Σουδάν και Νότια Αλγυρία στο νότο της Λιβύης βλέπουμε ότι έχουμε περιορισμένη ε, κρατική ε, εξουσία αυτών των χωρών. Δεν υπάρχει παρουσία κρατικών οργάνων και έτσι δημιουργήθηκε ένα κενό όπου αναπτύχθηκαν ε, τρομοκρατικές οργανώσεις. Πρέπει να φροντίσουμε ιδιαίτερα η εξαγωγή μικρών ελαφρών όπλων στην ε, ε, Αφρική να σταματήσει γιατί το πρόβλημα δεν είναι τα όπλα μαζικής καταστροφής αλλά ο ελαφρός οπλισμός που συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση πολλών κρατών. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Για δύο λεπτά τώρα το λόγο έχει η κυρία Δεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι σχεδόν συμφωνούμε σχετικά με την τραγικότητα της κατάστασης στο Μαλί. Εγώ θα ήθελα μόνο να ε, αναφέρω μία δυσφορία που αισθάνομαι απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί ε, έπρεπε να το είχαμε προβλέψει. Ήταν μία προαναγγελθήσα καταστροφή. Ε, διάφοροι συνάδελφοι που συμμετέχουμε στη δικασία και εδώ και μήνες από τότε που έχουμε την επέμβαση στη Λιβύη ε, μας λένε ότι κάτι κακό θα γίνει στο Μαλί. Το ακούσαμε και στο Τόγκο στην ε, συνεδρίαση με τις χώρες ΑΚΕ και την παραμονή του πραξικοπήματος ε, της Βρυξέλλες, ο συνάδελφός μας μας είπε μα, από το Μαλή μας είπε ότι μα, πρέπει να βοηθήσετε ε, επίκειται πραξικόπημα γιατί δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Είχαμε τη στρατηγική για το Σαχέλ, γνωρίζαμε τα πράγματα, ξέραμε ότι κάτι επρόκειτο να γίνει και σήμερα χαίρομαι που ακούω να λέτε ότι θα ε, πιέσουμε, ε, θα ε, επιδιώξουμε τον συντονισμό με τις γειτονικές χώρες θα ε, προωθήσουμε την ανάπτυξη, αναπτυξιακές δράσεις στις πιο φτωχές από τις περιοχές αυτές, αλλά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι νωρίτερα, ε, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι πρόκειται για μια πραγματική υπήρητη αποθήκη. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει νόημα να κλαίμε για το παρελθόν, να δούμε τι θα κάνουμε ε, από εδώ και πέρα. Όπως είπε όμως η κυρία Βερζιά, ήταν ένα πρόβλημα το οποίο ε, έβραζε και εμείς ε, ε, κατηληθήκαμε Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Συρνάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπος, ε, πολύ ε, δυσάρεστη η έκπληξη που έχουμε από το μαλή Έχουμε ε, ε, απαγωγές, ε, ε, αποσυνδικές τάσεις στον Βόρα, κίνδυνος διατροφικής κρίσης, προβλήματα που μπορούν να δηλητηριάσουν ολόκληρη την περιοχή. Το Μαλί όμως είναι μια παράπλευρη απολύτω, ένα παράπλευρο θύμα της σύγκρουσης στη Λιβύη. Ε, υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα το οποίο ξεπερνάει την πολιτική τάξη του Μαλή. Είναι ένα πρόβλημα που προέρχεται εκτός των σύνορων της χώρας, συνδέεται με το πρόβλημα της Λιβύης αλλά και ε, ευρύτερα με τα προβλήματα της περιοχής. Ε, στα πλαίσια μιας στρατηγική μετά τον Καντάφη για την ε, περιοχή αυτή χρειάζεται μια ε, πολιτική συνεργασία διότι θα πρέπει να βαθύνουμε στο πρόβλημα της ασφάλειας. θα πρέπει πέρα από τις επαφές που γίνονται με την ECOWAS ε, πρέπει και στη συνεργασία με τον ΟΗΕ να φροντίσουμε για ε, την ανθρωπιστική κατάσταση, γιατί όσο πιο καθυστερούμε, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η κατάσταση. Για ένα, για ένα λεπτό, κύριο Αλφόνση. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε τη Επιτροπή. ο λαός ε, του Τουαρέγ είναι περιθωριοποιημένος στην ευρύτερη περιοχή, στο Αζαγουάντ, το, την περιοχή των Τουαρέγ, του Τουαρέγ στο Μαλί, δόθηκαν πολλές υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν ποτέ. Γι' αυτό και το απελευθερωτικό κίνημα δίνει μάχη ώστε στο Σαγουάντ να αναγνωριστούν τα ιστορικά και πολιτιστικά και πολιτικά δικαιώματα των, ε, του ΑΡΕΚ. Είναι θεμητό. Βέβαια θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, να βελτιωθεί η κατάσταση, όχι να ε, ενισχύσουμε τους στρατιωτικούς για να καταπιέζουν τους του ΑΡΕΚ. Το απελευθερωτικό μέτωπο του Αζαουάτ δεν έχει καμία σχέση με τους Ισλαμιστές. Αντίθετα, ε, η Τουαρέκ είναι κατά της εφαρμογής ε, του Ισλαμικού νόμου της Αρία και έχουν ένα θυμικό δίκαιο πολύ πιο ανεκτικό απέναντι στις γυναίκες. Νομίζω ότι η ενίσχυση των Τουαρέγκ είναι καλύτερη εγγύηση κατά του Ισλαμισμού από ό,τι υποστήριξη των διαφόρων αυθαίρετων και αυταρχικών καθεστώτων. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και την αποκατάσταση τη σταθερότητα σε μια από τι πιο έθραυστε περιοχέ του κόσμου. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Κέλαμ. Ε, ε, κυρία, είπατε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ ειλικρινά για τα καθαρά και πιστικά σας λόγια για την κατάσταση στο Μαλί. Η εσωτερική σύγκρουση εκεί δείχνει πόσο έφραυστη είναι η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα σε εκείνη την περιοχή της Αφρικής. Επί 20 χρόνια το Μαλί παρουσιάζεται ως ένα πολυκομματικό, δικοματικό, ε, δημοκρατικό κράτος. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, ε, υπέστη πλήγμα η δημοκρατία και επί 11 ημέρες αποσχίστηκε το βόρειο τμήμα του Μαλή. Εκεί υπάρχουν στενές διασυνδέσεις με τρομοκράτες και με τους διαδόχους του Καντάφη. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε το ανθρωπιστικό πρόβλημα εκεί. Ε, ε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 1 δέκατο του πληθυσμού αντιμετωπίζει κατεπήγοντα προβλήματα και χρειάζεται τρόφιμα. Εκτός αυτού θα πρέπει να ε, υποστηρίξουμε αυτήν την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη χάρης στις μεγάλες προσπάθειες των αφρικανικών κρατών. Αν αποδειχθεί ε, θα πρέπει να ε, πείσουμε ότι δεν θα αποδεχθούμε στρατιωτικά πραξικοπήματα. Τότε υπάρχει ελπίδα για τη δημοκρατία. Όμως καταρχήν το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές αυτές, ούτως ώστε να μην υπάρξει ανθρωπιστική καταστροφή. Και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, όλοι ευελπιστούμε ότι η αποχώρηση των στρατιωτικών από την εξουσία θα θέσει τέρμα σε αυτή την αντιδημοκρατική παρένθεση στο Μαλί. Ελπίζω ο διορισμός του Πρόεδρου και του Πρωθυπουργού να θέσουν τέρμα σε αυτή την κρίση που μετά την στρατιωτική δικτατορία που ε, σταμάτησε το 2011 το 1991, συγγνώμη, ακολούθησε ένα δρόμο δημοκρατίας και σταθερότητας. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια τέτοια κατάσταση, να επαναφέρουν οι κάτοικοι του Μαρή τη δημοκρατία με ελεύθερες και ανώθευτες εκλογές. Επίσης θα πρέπει να διατρανώσουμε την υποστήριξή μας στην εδαφική καιρότητα του Μαλή. Η αποσχισμένη βόρεια περιοχή αντιμετωπίζει τη χειρότερη επιστηστική και ανθρωπιστική κρίση. Δεν θέλουμε ένα μαγκρέ που θα ελέγχουν οι εξτρεμιστές Ισλαμιστές. Δεν είναι για αυτό το λόγο που υποστήριξαμε την Αραβική Άνοιξη. Για 1,5 λεπτό το λόγο ο κύριος Φίσας Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βαρόνη, η τραγωδία του Μαλή είναι πραγματικά το χρονικό ενός προναγγελθέντος θανάτου. Πριν από ένα χρόνο είχα την τιμή να ε, είμαι επικεφαλής της ε, αποστολή παρατήρηση των εκλογών στον Νίγερα. Οι αρχέ του Νίγηρα που γνώριζαν πολύ καλά την κατάσταση ε, και ελάχιστοι πρέσβει ε, στην περιοχή αυτή έκλεισαν τον κόδωνα του κινδύνου στις, δημοκρατικές κυβερνήσει, στι ε, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τι τεράστιε και τρομέρε, επιπτώσει που θα είχε στην ζώνη Σαχέλ η επαναφορά των του που ανήκαν στου μισθοφόρους του στρατού του Καντάφη. Ήταν ένοπλοι του ΑΡΕΓ που θα επέστρεφαν και θα ενώνονταν με τους ομοθρίσκους τους και στις χώρες αυτές και στις δυνάμεις του Αλκίμη και μάλιστα ε, παρίσφρησαν και στις δυνάμεις του Ελκύμη μετά τις ανταρσίες που έγιναν στη Λιβύη. Όλα αυτά ήταν γνωστά, ε, γνωστές προειδοποίησεις ε, ε, από τους ε, εκπροσώπους της ζώνης Αχέλ. Θα πρέπει αμέσως να λάβουμε κάποια μέτρα, αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε ένα τραγικό πρόβλημα και πολύ, πολύ γρήγορα μπορούν, μπο, θα μπορέσουν οι χώρες αυτές να γίνουν ε, όμοιροι, έρμεα στα χέρια των δυνάμεων του Ακίμη και μάλιστα στα, προ, πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να απελευθερωθούν οι εχμάλωτοι και οι όμοιροι του Ακίμη, να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχουμε μόνο τον κύριο Φερέιρα στην, τον πρώτο ομιλητή. Ευχαριστώ οι εξελίξεις στο Μαλί επιδίνωσαν μια ανθρωπιστική κατάσταση που ήδη ήταν εξαιρετικά επισφαλής. Έχουμε μια όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια, επισητιστική απειλή με θάνατο και λιμοκτονία 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Έχουμε 200.000 πρόσφυγες στις γειτονικέ χώρες. Κρίσιμη κατάσταση στα σύνορα του Νίγηρα και της Μαυριτανίας. Όλες ε, οι πρόσφατες εξελίξεις είναι αναπόσπαστα δεμένες με την ε, ε, αθρώα εισρωή στο βόρειο Μαλί ε, όπλα που, από τη Λιβύη που είχαν εξαχθεί από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν στα, τη χώρα αυτή. Βέβαια, η ΕΚΟΒΑΣ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί μια διπλωματική και πολιτική διευθέτηση, χωρί όμω εξωτερικέ επεμβάσει και με την υποστήριξη του ε, τοπικού πληθυσμού και με σεβασμό τη κυριαρχία και τη εδαφική ακεραιότητα του Μαλή. Είναι τεράστια τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα τη χώρα. Ε, έχουμε θέματα επιστημικής ασφάλεια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε υγεία, διατροφή, κοινοφελεί υπηρεσίε. Η αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρουμε στη χώρα αυτή θα διαδραματίσει κέριο ρόλο. Σα ευχαριστώ. Δεν είχαμε άλλο μιλητή στο Catch the Θα ήθελα τώρα εν κατακλείδη να δώσω το λόγο για τα τελικά σχόλια στην Βαρόνια του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αξιότιμα μέλη για τα σχόλιά σας σχετικά με την εξέλιξη στο Ομαλή. Ε, σωστά είπατε ότι πρέπει να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν ζωτικά συμφέροντα για την ανάπτυξη της περιοχής. Ε, συλλογικές προσπάθειες χρειάζονται. Στενή επαφή και με τις γειτονικές χώρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολιτική αυτή μεταβατική φάση και βεβαίως ε, και στο... έχουμε την εμπειρία από την ακτή του Ελεφαντοστού και τις εμπειρίες ε, που είχαμε εκεί. Ε, παραμένουμε ανήσυχοι για την κατάσταση στο Βορρά και επαναλαμβάνουμε πάλι την υποστήριξή μας της εδαφικής ακεραιότητας του Μαλή. Ε, είμαστε σε επαφή με το ECOWAS για πολλά θέματα. Πώς θα συνεργαστούμε με αυτές τις ιδέες, πώς θα δημιουργήσουμε μια συλλογική δύναμη για να βοηθήσουμε την νόμιμη κυβέρνηση να αποκαταστήσει την τάξη σε όλη την επικράτεια. Επίσης ε, θα υπάρξει μια αποστολή πολιτική στα πλαίσια της πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας Επίσης ε, με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι πάρα πολλοί αναγκάστηκαν να διαφύγουν στο βορρά ε, στο μέσο μιας μεγάλης επισυδιστικής κρίσης. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ε, ανθρωπιστική υποστήριξη όπου μπορούμε λαμβάνοντας πάντα βέβαια υπόψη την σωματική ακαιρεότητα του προσωπικού μας και προσβλέπω στο ψήφισμα πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ για τα τελικά στους σχόλια. Έτσι τελειώνουμε το σημείο αυτό. Η ψηφοφορία για το θέμα αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης.